και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι τα πρακτικά της χθεσινής μας συνεδρίασης ε, διατίθενται ήδη. Ε, έχετε καθόλου ενστάσεις? Όχι. Ωραία. Άρα εγκρίνονται τα πρακτικά της χθεσινής μας συνεδρίασης.